Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ, έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη, το σχέδιο και το πρώτο σημείο σε αυτή είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, προτείνω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχετε κάποια αντίρρηση? Όχι. Εγκρίνατε επομένως. Σημείο 2. Όπως συνήθως Έχουμε την έγκριση των πρακτικών, των συνεδριάσεων μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Εφόσον πάλι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 10 η Ιουλίου και της 23 Ιουλίου. 23ης Ιουλίου. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Σημείο 3. Να σας ενημερώσω ότι έγινε συνεδρίαση των συντονιστών στις 18 Ιουλίου, όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν διαδικασίες της Επιτροπής μας. Τα πρακτικά της συνάντησης των συντονιστών, καθώς και οι αποφάσεις τους, βρίσκονται στους φακέλους σας. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με τα πρακτικά. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρίασης σήμερα, τα πρακτικά της συνεδρία των συντονιστών θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Σημείο 4. Ανακοινώσει του Προέδρου. Πολύ σύντομα σε αυτή τη φορά. Πρώτη ανακοίνωση λοιπόν, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μπορέσουν να μας δουν όσοι ενδιαφέρονται σε όλο τον κόσμο, από τη Λισαβόνα στο Λούνερπουργκ, από το Ταλίν στη Θεσσαλονίκη. Προσοχή λοιπόν, γιατί όλοι μας βλέπουν και μας ακούνε. Επίσης, υπάρχει διερμηνία Και για να μπορέσουν οι διερμηνείς να μεταφράσουν τα όσα λέτε με ακρίβεια, σας παρακαλώ να μιλάτε αργά και καθαρά έτσι ώστε να μπορέσουν. Αυτά τα δύο σύντομα θέματα κάτω από τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου και θα περάσουμε στο σημείο 5 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020. Εμείς ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου πρέπει να συζητήσουμε για την δική μας συνεισφορά και τις δικές μας αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Πρότεινα να μην συνταχθεί έκθεση, αλλά να στείλουμε μία επιστολή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, όπου θα κάνουμε ορισμένες τροπολογίες σε αυτόν. Μετά από συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες, καταλήξαμε σε υποβολή τεσσάρων μονοτροπολογιών, τρεις από τις οποίες είναι δικές μου και σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αύξηση ικανοτήτων, για τη δημιουργία ε, εργαστηρίων σχετικά με την κοινή διάσκεψη για τον ΠΟΕ. Ελπίζω να συμφωνήσετε με τις τροπολογίες αυτές και σε ό,τι αφορά το σχέδιο της επιστολής να σας ενημερώσω ότι όλες οι ομάδες συμμετείχαν στη σύνταξή της. και έχουν καταλήξει σε έναν συμβιβασμό, ο οποίο νομίζω ότι λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα όλων των πολιτικών ομάδων. Φυσικά, κάθε σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο, όπως και προτάσεις για διορθώσεις. Ε, και θα προσπαθήσουμε με τη σειρά μας να τις συμπεριλάβουμε στην επιστολή. Αυτά λοιπόν από εμένα και τώρα ο λόγος σε εσάς. Ποιο θέλει να μιλήσει για την επιστολή και για τι τέσσερι τροπολογίε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ω ΕΛΚ μπορούμε να στηρίξουμε την επιστολή ω έχει. Κάθε σχόλιο και κάθε μικρή τροποποίηση ελήφθη υπόψη. Φυσικά και υπήρξαν συμβιβασμοί. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκε και όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν σκληρά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εμείς στηρίζουμε τις πρώτες τρεις τροπολογίες απόλυτα. Σε ό,τι αφορά την τέταρτη από τον κύριο Σούλτς, θα μπορούσαμε να τη στηρίξουμε εφόσον δεχτεί να μειωθούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Πόζοα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα ECR μπορεί να στηρίξει το συμβαστικό κείμενο με μορφή επιστολής. Θα ήθελα όμως να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα που θα έχει ένα σκληρό άτακτο Brexit στην οποία περίπτωση θα είναι αναγκαίο να ληφθούν δημοσιονομικά μέτρα για την εφαρμογή του σεναρίου No Deal αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Χρειάζεται λοιπόν να ληφθεί υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος στην ευημερία και την απασχόληση των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν να τονίσουμε αυτήν την πιθανότητα και να ληφθεί υπόψη στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο δηλαδή, ένα άτακτο Brexit, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι δημοσιονομικά για το επόμενο έτος. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο συνάδελφο το λόγο. Α, όχι, εσεί κύριε Σόλτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και Σε ό,τι αφορά το σχόλιο του ΕΛΚ για την πρότασή μας σχετικά με τα νούμερα που έχουμε προτείνει. Προσπαθούμε με να ακολουθήσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τα ποσά, όμως θα επιμείνω. Χρειάζεται οι συμβουλευτικές ομάδες να έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το διάλογο και από τις δύο πλευρές και με την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να έρθουν σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το στάδιο της εφαρμογής, τα πέντε δηλαδή χρόνια που θα χρειαστούν. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα της διαδικασίας και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αρκετή στήριξη από τα κρατη Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και να εφαρμόσουμε τα δέοντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιστολή. Ε, με λυπούν λίγο τα σχόλια για το ότι κάποιες προτάσεις μας δεν συμπεριληφθήκαν πλήρως. Θα χρειαστεί να υπάρξει κάποια σύνδεση μεταξύ των ε, συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα μεταξύ των πολιτών, σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα, εμπορική πολιτική και πολιτική απασχόλησης, δηλαδή το πρώτο, μας, ε, το πρώτο σημείο. Εδώ θα θέλαμε να είχε ληφθεί υπόψη η διατύπωση που είχαμε προτείνει, δηλαδή η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας είναι πριν την εφαρμογή της και έπειτα χρειάζεται να γίνουν διεθνείς διασκέψεις έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις είτε υπό την αιγύδα των Ηνωμένων είτε διαφορετικά. Ευχαριστώ. Δέχομαι το σχόλιο σας και τη λύπη σας, όμως πολύ φοβάμαι πως τώρα πλέον δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Σοφία Μουνιάς από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους εσάς για την σύνταξη της επιστολής στην Επιτροπή Προϋπολογισμών η οποία επιστολή περιέχει όλες τις προτεραιότητες μας για την ε, εμπορική πολιτική. Θέλουμε να στηρίξουμε την mm. πολιτική αυτή με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελευταία ερώτηση, δηλαδή τη στήριξη που θα δώσουμε στην εφαρμογή του, των διτάξεων για το κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη και του περιβάλλοντος, να πω ότι αυτό είναι ένας τομέα στον οποίο στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε, όχι μόνο μέσω του επιχειρησιακού προπολογισμού τη Γενικής Διεύθυνση, αλλά και με άλλους τρόπους, με εξωτερικούς μηχανισμούς, για παράδειγμα. Έργο μας, λοιπόν, και καθήκον μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ε, συμβουλευτικές επιτροπές και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο τη ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το στηρίξουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Όπω σα είπα, εν μέρη μέσω του επιχειρησιακού προπολογισμού μα, αλλά και μέσω διαφόρων μέσων αποτρεπτικών. Όπως ε, έχει ακουστεί και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, η Επιτροπή σας θα εστιάσει όχι μόνο στο σχέδιο προϋπολογισμού που αφορά τις δικές μας επιχειρησικές δυνατότητες, αλλά στη χρηματοδότηση που μπορούμε να λάβουμε γενικότερα έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς με τη σειρά μας να εστιάσουμε στις δικές μας προτεραιότητες, οι οποίες είναι και δικές σας. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιστολή καλύπτει τις προτεραιότητες της ε, γενικής μας διεύθυνσης, η οποία έχει έναν μικρό μεν προϋπολογισμό, αλλά θα συνεχίσει να τον διαθέτει σε διάφορες ε, δραστηριότητες και μέσα που θα μας ε, βοηθήσουν να στηρίξουμε την πρόσβαση στην αγορά, την επιβολή και εφαρμογή της συμφωνίας, αλλά και την εφαρμογή της στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Μέχρι τώρα έχουμε στηρίξει όλες τις σχετικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν για την τροπολογία 4, το ποσό είναι ένα ποσό που σας βρίσκει σύμφωνο, κύριε Σόλης. Θέλετε απλά να, το αναφέρουμε ως ποσό ή... Νομίζω πως η πρότασή μας, την οποία στείλαμε στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών και την έχετε λάβει, αφορά δραστηριότητες οι οποίες ε, χρηματοδοτούνται από άλλη γραμμή του προϋπολογισμού. Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αν θα στηρίξουμε μια τέτοια πρόταση ή όχι. Η πρότασή μας παραμένει ίδια με εκείνη που υποβάλαμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Βέβαια, αν η Επιτροπή Προϋπολογισμών θεωρήσει ότι αυτό είναι προτεραιότητα και πώς χρειάζονται πρόσθετα κονδύλια για το σκοπό αυτό, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να στήσουμε κάποια project σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Τι συμπεραίνετε από όλα αυτά που ακούσατε για το συνολικό ποσό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ωραία, να προτείνω τότε να αυξήσουμε το ποσό και ελπίζω το ΕΛΚ να συμφωνήσει μαζί μου. Διότι θεωρώ πως χρειάζεται αύξηση. Έχει ήδη γίνει τέτοια ε, συζήτηση για το μέσο ε, που αφορά τις εταιρικές σχέσεις διότι δεν θα μείνουν κονδύλια καθόλου με την παρούσα σύσταση. Νομίζω πως το σκεπτικό μας είναι το ίδιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως χρειάζεται να υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια, τα οποία θα στηρίξουν τις ε, ομάδες αυτές, τις εγχώριες συμβουλευτικές επιτροπές. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μου για το ΕΛΚ. Να συμφωνήσουν δηλαδή για μία αύξηση του ποσού. Ωραία. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απορρίπτει την πρόταση για αύξηση, αλλά τώρα ο Χέλμουντ πρότεινε μία αύξηση κατά το ίμιση. Τι έχει να πει το ΕΛΚ. Το ΕΛΚ θέλει να κινηθεί στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής και δεν επιθυμεί αύξηση. Ωραία. Κάποιο άλλο σχόλιο. Κανείς. Θα ψηφίσουμε λοιπόν. Ο Χέλμουντ θα υποβάλει προφορική τροπολογία αύριο πριν την ψηφοφορία έτσι ώστε να γίνει αυτή η αύξηση και θα την ψηφίσουμε. Πολύ ωραία. Η ψηφοφορία λοιπόν θα γίνει αύριο στις 10 το πρωί. Αυτό θα γίνει και κλεισμένο των θυρών όπως και το σημείο παριθμών 7. Οπότε, παρακαλώ, Αυτοί οι οποίοι δεν επιτρέπεται να παρήνεται σε συνεδριάσεις ε, και κλεισμένο να εγκατέλειψουν το δωμάτιο και γι' αυτό